κατά την οποία θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Βλέπετε τους συναδέλφους από την Ουκρανία στις οθόνες σας. Meine Damen Κυρίες και κύριοι, μπορεί να υπάρξει κάποια καθυστέρηση κατά την μετάδοση. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό που λέμε εμείς εδώ μπορεί να καθυστερήσει 30 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό για να φτάσει στο Κίεβο και αντιστρόφως. Εάν στο τέλος της εισαγωγής μου λοιπόν μπορείτε να χειροκροτήσετε 30 δευτερόλεπτα θα μπορέσουμε να καλύψουμε την καθυστέρηση. Έχετε λοιπόν μια φορά επιτέλους ε, κάθε λόγο να χειροκροτήσετε. Κυρίες και κύριοι. Μετά θα περάσουμε στα διαδικαστικά που θέλετε να θέσετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε Ποροσέγκα, κυρίες και κύριοι, δεν υπερβάλλω πιστεύω όταν ε, θεωρώ ότι είναι ιστορική αυτή η στιγμή αυτή τη στιγμή εδώ το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και η Βερκόβνα Ράντα στο Κίεβο θα επικυρώσουν τη συμφωνία σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. Τα δύο κοινοβούλια ελεύθερα αποφάσισαν να κάνουν την ίδια χρονική στιγμή αυτήν την ψηφοφορία για αυτήν την συμφωνία. Αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία, ελεύθερα να αποφασίζουν τα κοινοβούλια, είναι το αντίθετο της χειραγωγούμενης δημοκρατίας. Η επικύρωση Κυρίες και κύριοι, η επικύρωση αυτής της συμφωνίας που έχει παραμείνει αμετάβλητη από τις πρώτες μέρες των ελεύθερων και ειρηνικών διαδηλώσεων στο Μάινταν είναι κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας με βάση αυτά τα οποία χρειάστηκε να δούμε τους τελευταίους μήνες. Ακριβώς θεωρούμε ότι ισχύει αυτό. Ποιο θα μπορούσε πριν από μερικά χρόνια, μερικού μήνε, να θεωρήσει ότι στην Ευρώπη θα τροποποιούνταν τα σύνορα μέσω άσκηση βία, ότι η ασφάλεια και η δομή ασφάλεια που φτιάξαμε στην Ευρώπη με τόσε προσπάθειε, ιδιαίτερα μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου, ποιο θα θεωρούσε πω είναι δυνατόν ότι θα μπορούσε να τεθεί ένα αμφιβόλο. Ποιο θα μπορούσε να θεωρήσει ότι το δίκαιο του ισχυρότερου για άλλη μια φορά θα ε, αντικαταστήσει στην Ευρώπη την ισχύ του δικαίου. Ο φόβο για την Ευρώπη είχε επανέλθει, ο για πολέμου είχε επανέλθει στην Ευρώπη. Αυτό που συμβαίνει στην ε, Ουκρανία και αυτό που συνέβη μα αφορά όλου. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Και τώρα που είμαστε σε σύνδεση με τους συναδέλφους στο Κίεβο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπερασπιστεί πάντα την εδαφική ακαιρεότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας. Πάντα το κάναμε στο παρελθόν και το κάνουμε και στο μέλλον. Και θα το κάνουμε αυτό ούτω ώστε ο λαός της Ουκρανίας που πολέμησε στο Μαϊντάν και είχε ένα όνειρο να μπορέσει αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Αγωνιζόμαστε για μια δημοκρατική Ουκρανία, κράτος δικαίου που να αναθεωρήσει τη σταγματική τάξη μια χώρα που θα εξαλείψει την διαφθορά, όπου θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάνω απ' όλα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων θα προστατεύονται υποστηρίζουμε μια Ουκρανία με ευημερούσα οικονομία, όπου θα κλείσει το κοινωνικό χάσμα και όπου όλοι θα έχουν ένα καλό μέλλον. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μάλλον όταν αυτό το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, αυτή τη μέρα η Ουκρανία θα έχει εκπληρώσει την υπόσχεση των ελληνικών διαδηλώσεων στο Μαϊντάν. Και νομίζω ότι εκφράζω την άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων όταν λέω ότι θα υποστηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό να εκπληρώσει αυτό το όνειρο του Μαϊντάν. Γι' αυτό γίνεται σήμερα αυτή η ψηφοφορία. Πριν τώρα περάσουμε στην ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία που γεφυρώνει τις αποστάσεις, να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσέγκα, ο οποίος θα μας μιλήσει από το Κίεβο. Και κατόπιν θα λάβει χώρα η ψηφοφορία και μετά την ψηφοφορία εγώ εδώ ενώπιόν σας θα υπογράψω την συνοδευτική επιστολή του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, ούτως ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της τελικής επικύρωσης. Και δίνω το λόγο τώρα στον πρόεδρο της Ουκρανίας, κύριο Παρασένκα. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε, πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόεδρε Σούλτς. Αγαπητέ Πρόεδρε Σούλτς, συμπολίτες Ουκρανοί, σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, πρώτα απ' όλα Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα χειροκροτήματά σας και για την στήριξή σας προς την Ουκρανία. Θέλω να σας πω ότι το κλίμα που επικρατεί εδώ, στην Βουλή, μου υπενθυμίζει πάρα πολύ την, το κλίμα που είχαμε εδώ και το 1991, όταν καταφέραμε να πετύχουμε την ανεξαρτησία μας. Κηρύξαμε την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ποιος είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του για την Ευρώπη. Αυτό είναι και το ζήτημα το οποίο θέτουν οι ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν να δούνε πώς επηρεάζει η Ευρώπη την κατάσταση στη χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσικό να δίνει κανείς τη ζωή του και να χάνει και τη ζωή του για τη χώρα του. Οι πρώτοι 100 Ουκρανοί που έχασαν τη ζωή τους τον Φεβρουάριο και οι υπόλοιποι που έχασαν τη ζωή τους στον ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας έχασαν τη ζωή τους όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά για τη θέση της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κανένα άλλο έθνος δεν τιμήθηκε τόσο πολύ και δεν πλήρωσε τόσο μεγάλο τίμημα μάλλον για την επιθυμία του να συμμετέχει στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πείτε μου, ποιος θα κλείσει, θα τολμήσει να κλείσει την πόρτα της Ευρώπης στην Ουκρανία, ποιος θα μπορούσε να είναι κατά της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είναι ο στόχος μας και σήμερα παίρνουμε το πρώτο βήμα, κάνουμε το πρώτο βήμα που είναι τόσο αποφασιστικής ε, σημασίας. Εφτά χρόνια μετά από τη διάσκεψη του Παρισιού ετοιμάσαμε το κείμενο αυτό της Συμφωνίας Σύνδεσης. Και θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχατε στη διαδικασία αυτή, τους διπλωμάτες πρώτα απ' όλα, τους εμπειρογνώμονες, αλλά και βέβαια πάνω απ' όλα τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι με αποφασιστικότητα στήριξαν την πορεία αυτή. Το φθινόπωρο που μας πέρασε είχαμε την εντύπωση ότι ήταν όλα έτοιμα για την υπογραφή, γιατί ολόκληρη η χώρα ήταν υπέρ της συμφωνίας αυτής. Τα επιχειρήματα αυτών που ήταν κατά ήταν πάρα πολύ αδύναμα. Όμως στις 29 Νοεμβρίου στο Βίλνιους όταν όλοι περιμέναμε την συμφωνία αυτή, την υπογραφή της δηλαδή, και όλοι αναφερόμαστε στην αναγκαιότητα υπογραφής αυτής της συμφωνίας, που ισχύει τότε όπως ισχύει και τώρα, οι Ουκρανοί αντέδρασαν στην ε, συμπεριφορά του Γιαννούκοβιτς, ο οποίος ε, τελικά θέλησε να μας στερήσει τη συμφωνία αυτή. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι η σημερινή μας ψηφοφορία θα αποδείξει ξεκάθαρα ότι όσες δυνάμεις μέσα και έξω θέλουν να σταματήσουν την πρόοδό μας έχουν ήδη ιτηθεί. Ξέρετε ότι η συμφωνία αυτή υπογράφηκε ήδη τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες και ταυτόχρονα επικυρώνεται σήμερα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για μας τους Ουκρανούς, αλλά για ολόκληρη την Ενωμένη Ευρώπη, γιατί χωρίς την Ουκρανία δεν υπάρχει Ενωμένη Ευρώπη. Εμείς δεν υποχωρήσαμε σε κανέναν εκβιασμό αντέξαμε. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι το κείμενο της συμφωνίας αυτής δεν έχει καμία παράγραφο, κανένα κόμμα, καμία λέξη που να πρέπει να αλλάχθεί. Αυτό το κείμενο λοιπόν θα υπογράψω και εγώ και θα επικυρώσω σήμερα. Ζητώ από την Ουκρανική κυβέρνηση αύριο να θέσει σε εφαρμογή τη συμφωνία αυτή. Αγαπητοί φίλοι, η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής είναι κάτι απλό. Πρόκειται για την ελευθερία λόγου, πρόκειται για κατάργηση θεωρήσεων, πρόκειται για τη δημοκρατία. Όλα αυτά είναι που θα βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε περισσότερο. Στις τελευταίες διαπραγματεύσεις που είχαμε στις Βρυξέλλες μπορέσαμε να διευρύνουμε ακόμα και αυτά που προβλέπει η ίδια η συμφωνία. Διακριτική μεταχείριση θα υπάρχει μέχρι το 2015. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα ε, μετά θα έρχονται στην δικιά μας αγορά στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Η Ουκρανία λοιπόν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί με άλλες χώρες, με άλλους παραγωγούς. Θέλω επίσης σήμερα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτήν την μεγάλη στήριξη που μας έχετε προσφέρει μάλιστα σε τόσο δύσκολους και περίπλοκους καιρούς. Οι εταίροι μας ένα πράγμα θέλουν σε αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις. Συνεπώς, μην καθυστερήσετε περισσότερο. Ούτε ο πόλεμος, ούτε η όλη κατάσταση μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την καθυστέρηση της συμφωνίας αυτής. Το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων για το 2020 να ξέρετε ότι θα υποβληθεί. Μαζί λοιπόν, χέρι-χέρι θα προχωρήσουμε. Δεν θα σκεφτόμαστε ο καθένα τον εαυτό του. Όχι, ο πρόεδρο, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, όλοι μαζί θα συνεργαστούμε και θα νικήσουμε στο τέλος. Αν κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει μέτωπο κατά των σχεδίων μας αυτών, θα αποτύχει. Οι μεταρρυθμίσεις προβλέπονται η Ουκρανία πρέπει να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό κέντρο αγώνα κατά της διαφθοράς. Εγώ θα προτείνω λοιπόν τέτοια νομοθεσία κατά της διαφθοράς στα πλαίσια της νομοθεσίας μας. Είναι κάτι που το αναλαμβάνουμε εμείς και το χρωστάμε στην επικύρωση και στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να πούμε ότι έχουμε ήδη αρχίσει την πορεία μας. Ένας ε, μεγάλος Ουκρανός συγγραφέας, ο Μιχάλης, είπε τον προηγούμενο αιώνα «Δώστε μας την Ευρώπη». Εμείς αντιλαμβανόμαστε την Ευρώπη σαν μια ψυχολογική κατηγορία η οποία μας επιτρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, στην πρόοδο. Σήμερα λοιπόν αυτό ακριβώς κάνουμε. Κάνουμε βήματα προς αυτήν ακριβώς την νέα κατεύθυνση, σε αυτόν τον νέο δρόμο επιστροφής μας στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά θα πετύχουμε. Ζήτω η Ουκρανία, ζήτω η Ευρώπη. Шановні колеги, нагадаю, що нам ще треба проголосувати. Це зараз буде просто історична мить, коли ми разом. Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για την Ουκρανία σήμερα. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν αποφασίζουμε. Με αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να προτείνω να ψηφίσουμε τώρα το νομοσχέδιο 0098 για την επικύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Πριν ψηφίσουμε όμως επιτρέψτε μου να σας πω τα εξής. Ποτέ στα χρονικά του κοινοβουλευτισμού δεν έχει υπάρξει παράλληλη ψηφοφορία δύο κοινοβουλίων που επικυρώνουν μια διεθνή σύμβαση. Ποτέ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι νομίζω μοναδικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός για το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι Ναι, ναι. Γι' αυτό κύριε και κύριοι, τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Οι συνάδελφοι είδαν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Κίεβο. Ξεκινάμε τώρα την διαδικασία ψηφοφορίας της Συμφωνίας Σύνδεσης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Είναι η έκθεση Σάρους Βόλσκι, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για να δούμε αν λειτουργεί και η δική μου κάρτα ψηφοφορίας. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Ψήφισαν 536 υπέρ, 127 ε, κατά και 35 αποχές. Κυρίε και κύριοι, όμω δεν ε, έληξε ακόμη ψηφοφορία. Χαίρομαι που είστε τόσο επιμελεί. Ψηφίσαμε την έκθεση Σάρου Βόλσκι. Τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση του συναδέλφου Μωράε για την περαιτέρω εξέταση των ε, μέτρων αυτών, ιδιαίτερα σε σχέση με του πολίτε τρίτων χωρών τη Σύμβαση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. ...539 υπέρ, 123 κατά, 33 αποχές. Και αυτή η έκθεση εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, είδατε ότι ο πρόεδρος Προσέγκο από την άλλη πλευρά ήδη έχει υπογράψει την θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Θα υπογράψω τώρα τη συνοδευτική επιστολή του Κοινοβουλίου που ενημερώνει τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης ότι εμείς επικυρώσαμε και καλούμε τα άλλα θεσμικά όργανα να θέσουν σε ισχύ αμέσως αυτή τη συμφωνία. Βεβαίω θα γίνει ενώπιον σα για να δείτε ότι συμβαίνει αμέσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Θέλει κανείς το λόγο. Όχι. Ωραία. Λίγη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Das sind Announcements, die ich jetzt mache, ne? Ist das Κυρίες και κύριοι, έχουμε μερικές ανακοινώσεις και τις επεξηγήσει ψήφου. Παρακαλώ όσους δεν θέλουν να συμμετάσχουν περαιτέρω στη διαδικασία να βγουν ταχαίως από την αίθουσα.